Euh, chers collègues, euh, merci de votre présence. Je propose que nous commencions nos travaux. Νομίζω ήρθε η ώρα να αρχίσουμε τις εργασίες στις συνεδριασίες μας. Ένας αριθμός συναδέλφων μας έχουν ήδη δηλώσει ότι κολλείονται σήμερα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον ε, αγαπητό Κέρμελ που είναι εισηγητής δύο σημαντικών θεμάτων τα οποία συζητεί επί του παρόντος η Επιτροπή Θεμελιωτών Ελευθεριών. Πρόκειται για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ σημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και επίσης το άλλο είναι για έλεγχο συνόρων και θεωρήσεις. Είναι βέβαια πολύ κοντά τα δύο θέματα. Ωστόσο, το ένα αναφέρεται σε θεωρήσεις και σύνορα και το άλλο σε συνεργασία αστυνομικών αρχών. Δίνω το λόγο στον κύριο Κέρμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω λίγο πολύ τα είπατε τα πιο σημαντικά και θα μπορούσα εγώ απλώς να βάλω μια τελεία. Αλλά παρόλα αυτά να δώσω λίγες λεπτομέρειες ε, στις και στους συναδέλφους. Ίσως θα πρέπει να σημειώσω πρώτα ότι πρόκειται και για εξυγχρονισμό ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και για συμπλήρωσή τους Κάθε ένας που γνωρίζει κάπως τα πράγματα στον χώρο αυτό γνωρίζει ότι κάπου αρχίζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, διότι κάποιος έρχεται και καταθέτει μια καλή ιδέα και μετά προκύπτουν λύσεις για κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Αλλού υπάρχουν ίσως διαφορετικές απαιτήσεις, κάποιος άλλος προτείνει κάποια άλλη λύση και έτσι τελικώς υπάρχουν καλά project με διαφορετικές όμως λύσεις και δεν είναι διαλειτουργικά. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή το σημείο διατομής όπως λένε οι ειδικοί για να μπορούν να συνδεθούν οι διάφορες αυτές λύσεις. Σε ό,τι αφορά δεδομένα προσώπων υπάρχει βέβαια και η έξτρα απέτηση ότι δεδομένα προσώπων πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο. Πρέπει ε, επίσης να γίνεται η διαχείρισή τους με ευαισθησία και επομένως και το επίπεδο ασφαλείας να είναι υψηλό. Εν ώψη αυτού κάνει πρόταση τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνοντας διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων να δημιουργηθεί ένα. Βεβαίως νομικά και τεχνικά θα διαχωρίζονται ώστε να είναι υψηλό το επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, να μην έχουμε αυτό που λένε ορισμένοι τον ε, διάφανο πολίτη. Βέβαια, η προτινόμενη λύση είναι σίγουρα η ιδεώδης, αλλά δεν θέλουμε ακριβώς να έχουμε κάπου αποθηκευμένα όλα τα ε, δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει εδώ χρειάζεται κάποια ε, ευαισθησία και κάποια προσοχή. Νομίζω πάντως ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ορθή εξακολουθεί δηλαδή να εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι ξεχωριστά, όμως υπάρχουν όπως είπα σημεία διατομής, τα οποία σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να συνδεθούν τα συστήματα αυτά ώστε να χρησιμοποιηθούν όπως προβλέπει ο νόμος. Πρόκειται τώρα για την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια καλύτερη διασυνδεσιμότητα. Εδώ αυτό φέρει τον τίτλο διαλειτουργικότητα. Αυτήν προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε για διαφόρους τομείς και ιδίω για το CIS, δηλαδή το SIS μάλλον, το σύστημα πληροφοριών Schengen, το Eurodac, το σύστημα πληροφοριών προξενικών θεωρήσεων, Visa, και τρία νέα πρόσθετα συστήματα, το σύστημα εισόδου-εξόδου, το λένε αυτό στα αγγλικά EES, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αδειών Ταξιδίου, έτιας, και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόριων Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών που έχει τα αρχικά έγκριση και το οποίο έχουμε συζητήσει προ λίγων μηνών. Για να συνδεθούν αυτά, θέλουν να φτιάξουν μια πύλη αναζήτησης, ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την σύγκριση και ανταλλαγή βιομετρικών δεδομένων και ένα detector για διάφορα στοιχεία ταυτότητας. Αυτά είναι αναγκαία για να αποφευθεί ώστε πρόσωπα με ψευδόνυμα ή δηλώνοντας ψευδή ονόματα να, είναι μεν, να περιέχονται μεν στην ε, τράπεζα δεδομένων, να μην μπορούν όμως να κάνουν οι αρχές ανταλλαγή δεδομένων και να βρουν ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν τώρα ευφυή μυαλά τα οποία έχουν προτείνει λύσεις για βελτίωση τουλάχιστον. Και Κοιτάξτε, ένα αμφιβολία θα πρέπει να δεχθούμε την πρότασή τους, διότι πρόκειται για εξαιρετικά τεχνικές λεπτομέρειες που τουλάχιστον εμένα ξεφεύγουν από τον ελεγχό μου. Και τα πράγματα αυτά που προτείνει η Επιτροπή φαίνονται λογικά και είμαι βέβαιος ότι είναι κιόλα. Για την προστασία δεδομένων είπα ήδη κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να εμβαθύνω, άρα πρόκειται περί του ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τράπεζες δεδομένων Interpol και Europol, θέλουμε να διασυνδεθούν. Επίσης θέλουμε ό,τι υφίσταται σε εθνικό επίπεδο να ενταχθεί και αυτό σε αυτήν την διαλειτουργικότητα. Πιο συγκεκριμένα, για τον δικό μας προϋπολογισμό, τα πράγματα αυτά σημαίνουν ότι αυτές οι τέσσερις συνιστώσεις διαλειτουργικότητας και η κεντρική αποθήκευση όλων αυτών των δεδομένων πρέπει να δημιουργηθούν και πρέπει να ε, είναι λειτουργικά. Επομένως πρέπει να γίνει ε, η μετακίνηση των δεδομένων, να εξασφαλιστεί η λειτουργία των σημείων διατομής και βέβαια πρέπει να εκπαιδευτεί και το προσωπικό. 424 εκατομμύρια κόστος για τα έτη 2019 έως 2027, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια ανά έτος. 25 εκατομμύρια για τον EU Lisa, μηχανισμό EU Lisa, 136 για αλλαγές στις χώρες μέλη, εκατομμύρια, 49 εκατομμύρια για την Ευρωπόλ και τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρονικών του συστημάτων, 5 εκατομμύρια ευρώ για τον οργανισμό Frontex, 2 εκατομμύρια ευρώ για την ΣΕΠΟΛ, που πρόκειται για οργανισμό που φροντίζει για την εκπαίδευση, και περίπου 8 εκατομμύρια για την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών της Κομισιόν. Αυτά φτάνουν τα 424 εκατομμύρια ευρώ και το πιο σημαντικό είναι 225 εκατομμύρια ευρώ για τον EU χωρίζεται σε 68 εκατομμύρια για την ανάπτυξη του συστήματος, 56 έξοδα διατήρησης, συντηρησής μάλλον, για την migration των δεδομένων 25 εκατομμύρια και 19 εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό και προσαρμογή του συστήματος έγκρισης. Είναι σημαντικό το έργο και από άποψη ύψους επενδύσεως. Θεωρώ όμως ότι είναι ορθή η επένδυση αυτή. Πρόκειται για επένδυση η οποία ε, αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια στην Ευρώπη και προσφέρει και υψηλό επίπεδο ασφαλείας, προστασίας δηλαδή προσωπικών δεδομένων. Είμαι βέβαιο λοιπόν ότι εδώ ανταποκρινόμαστε στι επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή δίνουμε στις αρχές ασφαλείας την αναγκαία εργαλειοθήκη ώστε να μπορούν να εργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο. Κάτι το οποίο είναι επίσης αναγκαίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι θα αναλάβουν την εκτέλεση της υπόθεσης αυτής θα πρέπει να δείξουν πνεύμα εξοικονόμησης και αποτελεσματικότητας. Δηλαδή θέλουμε να μπορούμε να βασιζόμαστε στον υπολογισμό που έχει τεθεί υπόψη μας, να μην έρθουν να μας πούν στη διάρκεια του προγράμματος ότι δεν τους αρκούν οι προγραμματισμένες θέσεις προσωπικού για παράδειγμα και πρέπει να υπάρχει και υψηλή διαφάνεια του κόστους. Είπα αρχικά ότι μιλούμε για πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Αν κανείς δεν είναι ειδικό της πληροφορικής και εφόσον ασχολείται με το θέμα αυτό, αναγκαστικά είναι υποχρεωμένος να πιστέψει τι του λένε οι ειδικοί. Όμως, κατά την εκτέλεση των μέτρων θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις και τις προμήθειες θα υπάρχουν αρκετές προσφορές ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση και ότι για τα χρήματα που θα διαθέσει ο προπολογισμό θα λάβει επαρκή ανταπόδοση. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορώ να συστήσω στην Επιτροπή Προπολογισμών να υπερψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κιόλμελ, Θα δώσω το λόγο σκιώδη ε, ομιλητές. Ο κύριος Φερνάνδες από το ΕΛΚΑ, που αντικαθιστά τον κύριο Λαμασούρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αντικαταστήσω τον Αλά Λαμασούρ. Δεν είμαι τόσο ικανός ο εκείνος. Θα προσπαθήσω όμως. Ο κύριος Λαμασού, ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να έρθει. Ευχαριστεί τον εισηγητή για την ποιοτική δουλειά του. Για αυτά τα θέματα, ο Αλάν Λαμασούρ θεωρεί ότι είναι επίγον για την ασφάλεια της Ένωσης ε, και την ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης ε, και τη μετανάστευση. Ως κοιόδης εισηγητής, ο κ. Λαμασού είναι πολύ υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ποσά των πιστώσεων που προτείνονται. Θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Η Δημοσιονομική Αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τη λειτουργία των νέων εργαλείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουάρδια Θαβάλ, που αντικαθά την κυρία Ταπαλδέλ, η οποία δεν μπορεί να παραστεί επίση στην συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λιεντέλ. Όλοι αντικαθιστούμε κάποιους που λείπουν. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κιόλμελ για τις προτάσει του και επομένως σε ευχαριστώ που αναφέρθηκες αποκλειστικά και, στο, και αποκλειστικά στο τμήμα του προπολογισμού. Κάτι που θέλω να ρωτήσω την εισηγητή αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λέτε ότι αυτό θα καλυφθεί από το σημερινό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Γιατί υπάρχει, λέει, αρκετά υπάρχουν αρκετά λεφτά. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση καταρχήν. Γιατί ούτω ή άλλω δεν θέλουμε να περικόψουμε ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Ούτω ή άλλω ακριβώ αυτή είναι η ιδέα, η λειτουργία των προγραμμάτων. Ε, γι' αυτό υπάρχει για να γίνονται και τέτοιου τύπου χρηματοδοτήσει. Ε, πέστε μου, Πού οφείλεται αυτή η επάρκεια των πιστώσεων, ε, σε ποιο ύψος στάουν οι πιστώσεις του ταμείου αυτού κτλ. Επίσης, μήπως θα μπορούσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό που λέει το να περικόψουμε τις προθεσμίες από τον ένα χρόνο στους έξι μήνες μου φαίνεται λίγο υπερβολικό και πρόωρο να το πούμε, αλλά τέλος πάντων γενικά συμφωνώ με την έκθεση. Ευχαριστώ. Έντερ. Λοιπόν, εγώ είμαι ο σκιώδης ηγητής της ομάδας των φιλελεύθερων. Είμαι και μέλος Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα σεβαστώ αυτό που είπε η Έντερ και θα αναφερθώ. Ε, πρόκειται για στρατηγικής σημασίας θέμα. Έχουμε διάφορα πληροφοριακά συστήματα κεντρικά που δεν έχουν καμία διασύνδεση μεταξύ τους. Έχετε το Schengen, το SIS δηλαδή, έχετε το VIS, το σύστημα για τις θεωρήσεις, έχετε το Eurodac για, τα, για τους υπηκόους που διαμένουν παρατύπω στο καλύτερη δυνατή. Και αυτό χρειάζεται για την ασφάλεια των συστημάτων και των έλεγχων της μετανάστευσης. Τούτου λεχθέντος, ευχαριστώ τον εισηγητή. Πάντως, θα ήθελα να του πω ότι υπενήχθηκε ότι ορισμένα στοιχεία του νέου συστήματος διαλειτουργικότητας τα κράτη-μέλη θα θεωρήσουν ότι χρειάζεται ένα backup, δηλαδή ένα σύστημα ασφάλειας ε, το οποίο θα έχει ένα κόστος. Ας τα πλαίσια λοιπόν των διαπραγματεύσεων που θα γίνει μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου υπάρχει συμφωνία που θα είναι ποιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρχει προς αύξηση του κόστους λοιπόν εκεί κατά πάσα πιθανότητα. Του του υποστήριζω και εγώ την έκθεση του Κέλμεν. Η κυρία Γκουάρδια Θαβάλ έθεσε ένα ερώτημα ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσε να απαντήσει η Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξη που δίνει στην πρόταση της Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη και να μισιώνω ότι τα προγράμματα θα πρέπει να είναι να ολοκληρώνονται με καλή σχέση κόστους αποτελεσματικότητας. Σε ό,τι αφορά το, θέμα της, το ερώτημα της κυρίας Γκλωρία Θαβάλ, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 2019 και το 20 είναι 32 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από το 10% του συνόλου. Το 2019 και το 20 είναι 32 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από το 10% του συνόλου. 32. Αυτά τα 32 θα πρέπει να τα βρούμε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τώρα, για την συχνότητα υποβολής εκθέσεων Η Κομισιόν συμφωνεί μαζί σας και θα ήθελα να υπενθυμίσει ότι ο κανονισμός για το σύστημα εισόδου-εξόδου τέθηκε σε ισχύ τέλη του περασμένου έτους. Σε αυτόν τον κανονισμό, στην τελική εκδοχή που υιοθετήθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για το Ιουλί, για αυτό το πρόγραμμα διαλειτουργικότητας. Δύσκολη λέξη, την περδεύω λιγάκι μερικές φορές που συζητάμε σήμερα. Από πλευράς Κομισιόν, λοιπόν, οι τροπολογίες που προτάθηκαν μέσω του 237, το πρόγραμμα διαλειτουργικότητας είναι λιγότερο επικίνδυνο από το πρόγραμμα εισόδου-εξόδου. Επομένως, θα ζητούσαμε να μην ζητήσετε από εμά μεγαλύτερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων πέρα από αυτές που ήδη προτείναμε εμείς. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Καταγράψαμε την πρότασή σας, αλλά εμείς αποφασίζουμε βεβαίω. Μιλάμε για την ε, δική μας Επιτροπή, έτσι, την Επιτροπή Προπολογισμών. Ο κ. Χάουαρθ τώρα θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο οι τεχνολογίες διατελειτουργικότητας ε, ε, διτύφονται εδώ και κάποιο όλο το ζήτημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω εξή προ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό έχει κλείσει μια χρόνια, βλέπω. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ε, κίνδυνο που προκύπτει από κάποιες τεχνολογίες. Προφανώς έχουν προωθήσει λοιπόν πώς θα γίνει η αξιολόγηση του κινδύνου και τι συνέπειες θα έχει αυτό για την χρηματοδότηση. Είναι ίσως δύσκολη αυτή η ερώτηση, αλλά φαντάζομαι ότι το σύστημα αυτό είναι απαραίτητο για την ε, δυνατότητα εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου των συνόρων. Και ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η περίοδος. ευχαριστώ κύριε Χάουαρτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει μήπως. Ναι, ευχαριστώ κύριε Διπρέ Για την ερώτηση αυτή θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο, ο οποίο είναι και υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Ο προπολογισμό ε, έχει βάση 9 ετών για να έχουμε μια ιδέα για το κόστος ως μακροπρόθεσμα, αλλά ε, ουσιαστικά η περίοδος αυτή και το κόστος είναι πολύ πιο μικρό σε ό,τι αφορά βραχυπρόθεσμα. Κοιτάξτε λοιπόν για το κόστος ως μακροπρόθεσμα, αλλά ε, ουσιαστικά η περίοδος αυτή και το κόστος είναι πολύ πιο μικρό σε ό,τι αφορά βραχυπρόθεσμα. Κοιτάξτε λοιπόν τα σχετικά έγγραφα. Θα δείτε ότι στη σελίδα 82 έχετε μια επισκόπηση για τα ποσοστά συντηρήσει αυτών. Σωστά φυσικά επισημάνατε ότι ενδεχομένως να υπάρχει εξέλιξη της τεχνολογίας σε τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι προφανώς εγγενές για όλα τα προγράμματα IT. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα μεταξελιχθούν στο σύστημα πληροφόρησης ε, θεωρήσεων. Το ίδιο συνέβη. Αλλά μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί, εξελέχθηκε. Εξελέχθηκε το σύστημα προφανώς και χρειάστηκε ανάλογη χρηματοδότηση. Άρα όλοι ουσιαστικά εργαζόμαστε βάσει των... Ο κύριος Χάουαρ θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, όχι, ευχαριστώ πρόεδρε. Μάλιστα. Κανείς άλλος θα ζήτησε το λόγο και γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μας, τον κύριο Κολμέλ, για να κάνει τα καταλητικά σχόλια σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους έτσι. Θα παρακαλέσω τον κύριο Φερνάντες να τον, ο οποίος θα αντικαθιστά, ε, να ε, κάνει τη φορά την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για λογαριασμό της Air France. Ο εισηγητής μας είναι θετικός και απέναντι στο Ταμείο αλλά και στην κινητοποίησή του για το συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ και μια δεκαετία πολλοί κόσμος έχει ωφεληθεί από τις παρεμβάσεις του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι στις 8 έκτου 2017... Ότι θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα, αυτόν τον κανονισμό. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η Air France θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της ε, στο εσωτερικό και θα πρέπει να προβεί σε κοινωνικό διάλογο με τους εργαζομένους της. Κάτι που μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχει συμβεί, στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε να συμβεί. Και πρέπει να δούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στις, ε, και στην ε, Γαλλία, αλλά και στις ε, εταιρείες που κάνουν υπεργολαβίες για την Air Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα στο οποίο και διαπιστώνουμε εκ νέου ότι το Ταμείο αυτό προφανώς ε, έχει ε, πολλά, πάρα πολλά λόγοι όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπαρέμβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά τις αρμοδιότητες της αυτά είναι εθνικά καθήκοντα. Γιατί δάλλως θεωρώ ότι κάνουμε αυτό που μας ε, κατηγορούν οι πολίτες ότι κάνουμε ότι είμαστε αδιαφανείς και χρηματοδοτούμε μέσα από το Ταμείο Προσαρμογή στην Προκοσμιοποίηση πολύ διαφορετικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόλμπελα. Ο κύριος Περνάντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι οι απολυθέντες έχασαν δουλειά τους. Αυτό το ταμείο δεν έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό το σημείο. Εάν θεωρείτε ότι δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις εταιρείε. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματά σας, αλλά αυτό το ταμείο δεν δημιουργήθηκε για τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους. Δεν μας ενδιαφέρει από πού απολύθηκε. Από δημόσια εταιρεία, από ιδιωτική εταιρεία, από εταιρεία που έλαβε ευρωπαϊκή επιχορήγηση, επιδότηση. Είναι ένας άνθρωπος που έμεινε άνεργος ε, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε λοιπόν ένα ταμείο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε για να ξαναβρούν δουλειά. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο. Και για, ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες που χάσαν τη δουλειά τους. Μπορούμε να μην συμφωνούμε με τους κανόνες που υιοθετήθηκαν για το Ταμείο αυτό, αλλά εφόσον υιοθετήθηκαν θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει χρήση αυτού του ταμείου με σεβασμό των κανόνων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που απολύθηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κρέσλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι είναι περίεργη αυτή η αίτηση, αυτό το αίτημα. Είναι το δεύτερο αίτημα ουσιαστικά. Μα τη ίδια εταιρεία. Και μιλάμε και για μια εταιρεία η οποία 16% είναι στα χέρια της, ε, του γαλλικού κράτου. Νομίζω ότι ουσιαστικά ενθαρρύνουμε την Air France να συνεχίσει να κάνει τέτοια σφάλματα διαχειριστικά. αλλά πάρα πολύ αμφισβητήσιμο αυτό. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Α, Κιόλμελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εν συντομία για αυτά που είπε ο συναδέλφος ο κ. Φερνάντες η... το επιχείρημά του ότι εδώ μιλάμε για τους άνεργους και όχι για τις επιχειρήσεις ε, τυπικά στέκει αλλά δεν το εννοούσα καθόλου με αυτά που είπα και θα ήθελα να το διευκρινίσω δυστυχώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα 7% ποσοστό ανεργίας υπάρχουν κάποιοι κανόνες δεν λέω να με τηρούνται οι κανόνες, αλλά οι κανόνες αυτοί έχουν να κάνουν για κάποια πολλά, πολύ περιορισμένα φάλματα και κάποιες πολύ περιορισμένες περιπτώσεις από τα εκατομμύρια ανέργων. Άρα, αυτά που έχουμε ως σκοπό να κάνουμε με το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό και ζητείτε να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ασφάλεια για την ανεργία. Αλλά τότε θα είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των μεταφορών χρημάτων. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια λεπτομέρεια αν θέλετε, αλλά καταδεικνύει με σαφήνεια την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε και για τη διαφάνεια που επιθυμούμε. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε γιατί πάντα θα υπάρχουν ε, αν υπάρχουν ε, μάλλον ε, βουλευτές και ε, πολιτικές ομάδες που θέλουν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ασφάλεια για τους ανέργους, πολύ ωραία, έχουμε και εκλογές του χρόνου. Να βγουν, να το πούν ξεκάθαρα, να δούμε το θέλουν οι πολίτες ή όχι. Και μια προσθεκή εχθές, μιας και μιλήσαμε για θέματα χρηματοδότησης. Ίσως να ακούγεται πάρα πολύ σύγχρονο και πολύ αλληλέγγυο να λέμε ότι δεν κάνουμε πλέον διάκριση βάσει χωρών που είναι καθαροί εισφορείς καθαρή αλλά πρακτικά υπάρχει αυτή η καθαρη δικαιουχοι αλλα πρακτικα υπαρχει αυτη η διακριση και πολύ απλά όποιος... Ε, ευχαριστώ. Άκουσα αυτά τα σχόλια και δεν ξέρω αν ο κανονισμός για το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση στα γερμανικά σημαίνει κάτι άλλο. Εμεί δεν δίνουμε αυτά λεφτά για να διασώσουμε εταιρείε, σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους, βοηθάει τους εργαζόμενους που χάσαν τη δουλειά τους να κάνουν μια κατάρτιση ούτω ώστε να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασία. Ε, υπάρχει το, γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, ε, το έχουμε φτιάξει για εκείνους τους ε, Τώρα εσείς μιλάτε για αυτή την ευρωπαϊκή ασφάλεια για, τις, για την εργασία. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αν και εμείς οι σοσιαλιστές θα το θέλαμε, ας πούμε. Ε, θα το θέλαμε και ενώψη ευρωεκλογών και αν τα καταφέραμε μάλιστα θα ήταν πολύ θετικό να είχαμε μια τέτοια κάταξη της Επιτροπής μας, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό επίδομα ενεργείας. Εγώ δεν υπερασπίζομαι αυτό το ταμείο. Αν κοιτάξω την εκτέλεσή του, χρησιμοποιείται κυρίως για τις χώρες του Βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπερασπιστώ ε, την ιδέα ότι όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν ε, αυτό το ταμείο. Η Γερμανία το έχει χρησιμοποιήσει κατά επανάληψη. Το Βέλγιο επίσης. Η Φιλανδία πολλές φορές χρησιμοποιήσει το ταμείο. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε τη χρησιμοποίηση αυτό το ταμείου. Μπορείτε να το πείτε. Αλλά να το πείτε και στους Γερμανούς, οι οποίοι αποφελήθηκαν ήδη από το Ταμείο. Πρέπει να ξέρουν οι Γερμανοί ότι εσείς δεν θέλετε αυτό το Ταμείο. Δεν θέλετε αυτό το Ταμείο να υπάρχει για να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάσαν τη δουλειά τους. Αυτό το Ταμείο δεν είναι ένα Ταμείο υπέρ των επιχειρήσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αφορά τα άτομα. Τα άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους. Για να τα βοηθήσει για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι υπέρ των επιχειρήσεων αυτό το ταμείο. Νομίζω ότι αυτή είναι η σύγχυση από την οποία προκύπτουν και όλες αυτές οι παρεξηγήσεις. Τι Γκρέσλε, να σας πω και το εξή όμως. Σε ό,τι αφορά αυτό το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Θα έχετε, όσον ονούπο την ευκαιρία, να πείτε όλες αυτές τα επιχειρήματα. Γιατί πλησιάζει η προεκλογική εκστρατεία και κατά τη διάρκεια αυτή θα μπορέσετε να πείτε ενώπιον του κοινού όλε αυτέ τα, ιδέε αυτές και τα επιχειρήματα. Ε, εδώ θέλουμε... Πολύ ωραία. Οι ομάδες θα πάρουν θέση για το θέμα που μας απασχολεί, έτσι. Τα επιχειρήματα, αυτά θα τα αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Τελική ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Μιρεσάν για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2 στο γενικό προλογισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Όπω θα ξέρετε όλοι, αυτό ε, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού είναι. 2018 είναι αρκετά αυτοματοποιημένη αυτή η διαδικασία για μας. Το πλεόνασμα του περσινού Αμα έτος ήταν 545 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν εισαγάγουμε πλέον στον προϋπολογισμό του φετινού έτους και αυτό προφανώς θα μείωσε ασφαλώς να πάρουμε υπόψη τη συνολική εικόνα και το γεγονός ε, ότι πέρσι όπως είδαμε ότι ήταν ε, απογοητευτική η ε, υλοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεν πετύχαμε αυτά που περίμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάθηκε ταυτοτικός ε, προπολογισμό, ο υπαρχά θα κάναμε να μην ε, είμαστε περήφανοι ότι κάναμε φανταστική υλοποίηση του προπολογισμού πέρσι και να κοιτάξουμε μόνο τα 555 εκατομμύρια που είχαμε πλεόνασμα, να δούμε ποια είναι η συνολική εικόνα. Και να έχουμε υπόψη μας ότι το πλεόνασμα ήταν τόσο μικρό, ιδιαίτερα στο 1β, είχαμε ένα μεγάλο τμήμα των πόρων που δεν έφτασε στους δικαιούχους και γι' αυτό λοιπόν η υλοποίηση του προϋπολογισμού το 2018 είναι ακόμα πιο σημαντική και νομίζω ότι ο Πρόεδρος θα το συζητήσει αυτό στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2018 ότι πέρα από τα πλανάσματα αυτά τα οποία εισαγαγόνται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί εκ νέου έσοδα τα οποία προέκυψαν από πρόστιμα ή από καθυστερημένες πληρωμές χωρίς ε, μείωση όμως της συνεισφοράς βάση του ΕΧΠ από τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ανέκαθεν ναι, για μας. Και επίσης ε, με αυτό σχετίζεται και το εξή. η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού το οποίο θα ενταχθεί στα πλαίσια του προπολογισμού το οποίο σταδιακά και πρωτευτικά θα γεμίσει από απρόβλεπτα έσοδα, τα οποία και θα μεταφέρονται για να προβλέψουμε ακριβώς για απρόβλεπτα έξοδα. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο ως πολίτης ξέρω ότι κάθε ότι σε κάθε μήνα μάλλον πρέπει να έχω ένα ποσό στην άκρη για να προβλέψω για απρόβλεπτα έξοδα κάνουν κάποια αποταμίευση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην ε, κατάσταση των απρόβλεπτων έξοδων, αλλά δεν μας αφήνουν να κάνουμε καμία αποταμίευση για τα έξοδα αυτά. Θέλουμε να επιδείξουμε μια επιθυμιότητα. Λέμε ότι εφόσον υπάρχουν που υπάρχουν αυτά τα απρόβλεπτα έσοδα, αφήστε μας να τα αποταμιεύσουμε προκειμένου να έχουμε κάποια χρήματα όταν θα προκύψει ανάγκη. Και γι' αυτό λοιπόν στο Πουδοπού είδαμε πόσο σημαντικό ποσοστό ε, των έξοδων είναι τα πρόβλεπτα έξοδα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, τη δημοκρατία, τους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάτσουμε, να συζητήσουμε κατά πόσον ε, αυτή η διευκόλυνση για την Τουρκία θα συνεχίσει 3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά δεύτερον, παράταση του ΕΦΣΙ, του Προγράμματος Στρατηγικών Επενδύσεων, Έχουμε ιδέες και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πολλές, σε πολλές περιπτώσεις προσθέθηκαν πολλά τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα που δεν θα πρέπει φυσικά να διακυβεύουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα. Θα δούμε λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς θα αποταμιεύσουμε τα απρόβλεπτα έσοδα. Αυτά από πλευρά μου, Πρόεδρε. Αυτέ είναι οι πολιτικέ παρατηρήσει που είχα να κάνω και πιστεύω ότι είναι σημαντικά αυτά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε την ε, μελλοντική ε, υλοποίηση του προπολογισμού. Κατά τα άλλα, η άσκηση, όπω σα είπα, είναι αρκετά αυτοματοποιημένη. Έχουμε λοιπόν την έκθεση, το σχέδιο έκθεση με προθεσμία για καταβολή, υποβολή προθεσμιών ε, τροπολογιών, συγγνώμη, η 31η Μαΐου και θα ψηφίσουμε 18-19 Ιουνίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχει μιλήσει ο κ. Μουρεσάν. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκάρδια Σαβάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μουρεσάν. Για δύο λόγους. Αφενός το πλεόνασμα είναι μάλλον μικρό και έγιναν βέβαια οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί της ε, προηγούμενης χρονιάς, όπου φάνηκε καθαρά ότι ε, δεν έμε εάν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο. Το εξήγησε ήδη ο κ. Μωρισάν, δηλαδή να κάνουμε ένα αποθεματικό. Αν για παράδειγμα υπάρχουν επιβάλλονται χρηματικές ε, ποινές συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες στον να μπορούμε να αντιδράσουμε. Για παράδειγμα, με την, ε, για την ε, δήλωση με την Τουρκία. Εάν είχαμε το πρόνοσμα θα είχαμε και μια μεγαλύτερη ε, δυνατότητα να αντιδράσουμε. Και η θέση μας... Μια κουβέντα και εγώ, μιας και είμαι εδώ και ως φιλελεύθερος, συμφωνούμε και δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ήδη ο κύριος Μουρεσάν και η κυρία Γκαρδιά Ζαμπάλη. Συμφωνώ απολύτως με την ε, έκθεσή σας άλλωστε. Νομίζω ότι το οποίο να τροφοδοτείται από τα πρόστιμα και χρηματικέ ποινέ που επιβάλλονται στι επιχειρήσει. Και είναι κάτι το οποίο ζητούμε εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει και πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του νέου ιδίου πόρου που μπορούν να τεθούν στη διάθεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού Ωστόσο σε αυτή την πρόταση δεν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο αυτό. Εκφόλιεται σε δημοσιογικό πλαίσιο. Ο κ. Μουρεσάν σα εξήγησε πότε είναι και δυνατόν να κάνετε τροπολογίε με 31 Πέμπτου το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα τώρα τη ημερήσια διάταξη για το συγκεκριμένο σα υπενθυμίζω εάν έχετε λησμονήσει ότι ο πρόεδρο Αρτουή έχει αποστείλει επιστολή στην κυρία Καλβίνιο για ιδίω για, για τα αυτόνομα εμβάσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ορισμένες πιστώσεις και ορισμένες αποφάσεις που έχουν σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό, όπως για παράδειγμα η παράταση της ε, διευκόλυνσης προσφύγων με την Τουρκία. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία σχετικά με το οικονομικό έτος 2018 και μετά θα δώσω το λόγο πάλι στον Γενικό Εισηγητή κύριο Μου Ρεσάν. Εσεί, κύριε εκπρόσωπε τη ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχω να σας πω λίγα πράγματα. Πρώτα, εφιστώ την προσοχή σας στο νέο μορφότυπο της Weekly Implementation Report. Δεύτερο, δίνω μια συνολική εικόνα της ε, εκτέλεσης του προϋπολισμού. Τρίτο, για να είμαι πιο σαφή για την συνοχή ε, τίτλος 1β. Επίσης, σύντομη επισκόπηση των αυτόνομων εμβασμάτων. Πέμπτο, επανέρχομαι στις δεσμεύσεις για Συρία και Ιεμένη, όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή σας. Έκτο, σύντομη τοποθέτηση για το που βρισκόμαστε με τη διευκόνηση προσφύγων για την Τουρκία. Και τέλος, πού βρισκόμαστε με τους μελλοντικού διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Πρώτα, επισημαίνω στην Επιτροπή σας τη νέα παρουσίαση της Weekly Implementation Report, την οποία σας στέλνουμε στη τακτική βάση και που ελπίζω ότι επιτρέπει πλέον στα μέλη σας και στο προσωπικό σας να έχουν ταχύτερη κατανόηση για το πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός, διότι έχουμε βάλει, έχουμε εντάξει τις πληροφορίες ανά πρόγραμμα. Πολιτικά αυτό ε, καθιστά το πράγμα κατανοητότερο για τα μέλη σας. Επίσης, λόγω του ενδιαφέροντος που δείχνεται στις ε, αυτόνομες μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε δημιουργήσει δύο ξεχωριστές κατηγορίες στην έκθεση, αφενός μεταφορές της αρχής ε, προϋπολογισμού και άλλη για τις αυτόνομες μεταφορές πληρωμών. Μπορείτε να δείτε αμέσω δηλαδή αν έχετε μεταφέρει κάποια πιστώση μεταξύ προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν θέλετε μπορείτε να εξετάσετε και τι λεπτομέρειε μεταξύ των γραμμών του προπολογισμού. Ελπίζω να διεκτιμήσετε αυτό και ελπίζω να σα βοηθήσει στο έργο σα. Σε ό,τι αφορά τη συνολική εκτέλεση του προπολογισμού και σε ό,τι αφορά τι πιστώσει υποχρεώσεων για το σύνολο του προπολογισμού βρισκόμαστε στο 81% της εκτέλεσης Πέρσι στην ίδια περίοδο είχαμε φτάσει το 76%. Τα ποσοστά αυτά και φέτος και πέρσι είναι πολύ ψηλά. Και είναι λογικό αυτό διότι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες δαπανών, συνοχή και γεωργία, έχουν σχεδόν καλυφθεί πλήρω σε υποχρώσει πάντα βεβαίω, ε, πιστό υποχρώσαν. Είναι λογικό να είναι υψηλό το ποσοστό εκτελέσεων. Σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ, από σήμερα βρισκόμαστε σε επίπεδο εκτελέσεων 41%. Σε σύγκριση με πέρσι την ίδια εποχή ήμασταν στο 36% τότε μόνο. Άρα είμαστε κάπως καλύτερα από πέρσι, το οποίο εν πάση περιπτώσει καλό νέο είναι. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε ακόμα νωρί στο δημοσιονομικό έτος και είναι πρόωρο να συναγάγει κανείς αντίποτε συμπεράσματα για την ώρα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της εκτέλεσης στην συνοχή, πάντοτε για πληρωμές βέβαια, διότι βεβαίω οι υποχρεώση είναι πλήρης. Επιβεβαιώνω πρώτα ότι το μικρό αυτό και οι μικρές αυτές στερήσεις που είχαμε δει στο τέλος του 2017, 2,5 έως 3 δισεκατομμύρια νομίζω, αυτά καταβλήθηκαν αμέσως βέβαια με την αρχή του έτους, τον Ιανουάριο δηλαδή ήδη, και εκεί όπου βρισκόμαστε τώρα για φέτος είναι ότι από ένα προϋπολογισμό 47 δισεκατομμυρίων για πληρωμές στη συνοχή έχουμε εκτελέσει ως τώρα 7,5 δισεκατομμύρια. Θα έλεγα 16 με 17% του συνόλου. Οι νέες payment claims που έχουν λάβει οι χώρες μέλη για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους φτάνουν στα 5,5 δισεκατομμύρια. Πάλι αυτό είναι χαμηλό βέβαια ως ε, ποσόν στο σύνολο του προπολογισμού, αλλά δεν μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, διότι οι ίδιες οι προβλέψεις των χωρών μελών δείχνουν ότι θα υπάρχει ένα σημαντικό backlog, μια σημαντική υστέρηση στα τέλη του έτους. Όπως έγινε και πέρυσι λοιπόν μπορούμε να αναμένουμε ίσως το μισό, ίσως και περισσότερο από το μισό των ε, ε, αιτήσεων, των αξιώσεων να φτάνουν περί τα τέλη του Νοεμβρίου-Δεκέμβριο. Και αυτές οι νέες ε, πληρωμές που έχουν ζητηθεί έχουν καταβληθεί ή βρίσκονται στη φάση της καταβολής. Λόγω αυτού του backloading των προβλέψεων των χωρών μελών δεν θα μπορούμε να συναγάγουμε εύλογα συμπεράσματα για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στην συνοχή πριν από το τέλος Ιουλίου, όπου θα μας δώσουν ε, τις ε, ενημερωμένες προβλέψεις του μέλη και θα μας πούν αν διατηρούν τις προηγούμενες ε, προβλέψεις για το 2018 για τα payment claims ή αν έχουν κάνει προσαρμογές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όσον αφορά το επόμενο θέμα τώρα, τις αυτόματες τις αυτόνομες, συγγνώμη, τις αυτόνομες μεταφορές κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο ζητήματα εδώ στη συνοχή. Έχουμε μεταφέρει 45 εκατομμύρια μεταξύ κατηγοριών περιφερειών ως συνέπεια των, του αναπρογραμματισμού που κάνουν οι χώρες μέλη και μετακινούν κονδύλια ανάμεσα σε κατηγορίες περιφερειών και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να ακολουθήσει. Για τον τίτλο ή την κατηγορία 3 έχουμε μεταφέρει 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας στην Ευρωπόλ γιατί προέκυψε η την κατηγορια 3 εχουν μεταφερει 8 εκατομμυρια απο το ταμειο στηρικης ασφαλειας στην ευρωπολ χρηματοδοτήσεως για ικανότητες αποκρυπτογράφησης και να ενισχυθεί η Ευρωπόλ για δαπάνες που έγιναν με guest offices στα hot spot. Αυτές είναι οι αυτόνομες μεταφορές στις υποχρεώσεις τις οποίες θα θέσω υπόψη. Σε ό,τι αφορά τις αυτόνομες μεταφορές στις πληρωμές, κάνουμε πολλές τέτοιες, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία εντός προγραμμάτων εντός δηλαδή των κονδυλίων του προπολογισμού για συγκεκριμένα προγράμματα. Είναι επομένως περιορισμένη η σημασία τους για τα μέλη της Επιτροπής σας. Ό,τι αφορά κινήσεις πληρωμών μεταξύ προγραμμάτων ήταν εξαιρετικά περιορισμένες έως τώρα, όπως θα μπορέσετε να δείτε και στην εβδομαδία έκθεση. Τα ποσά είναι του 1 εκατομμυρίου, 1,5, 2 εκατομμυρίων, πολύ περιορισμένα ποσά. Δεν έχω δηλαδή τίποτα ιδιαίτερο να επισημάνω σε σας σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της Κομισιόν για Συρία και η Εμπένη, εδώ... ε, μου ζητήσατε να σας ε, ενημερώσω και θέλω να σας ενημερώσω πολύ σύντομα. σε ό,τι αφορά τη Συρία έχουμε στείλει γραπτή ενημέρωση στη γραμματεία της Επιτροπής σας με λεπτομέρειες για τις ε, δεσμεύσεις μας που έγιναν κατά τη διάρκεια τη διάσκεψης τον περασμένο μήνα 23 και 24 Απριλίου. Όπω και τα προηγούμενα χρόνια, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί έχει δεσ... να δώσει 560 εκατομμύρια ευρώ, ε, αυτό δεσμεύει βασικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχει μπει στο σχέδιο προπολογισμού του 2019 που θα υιοθετήσει η Κομισιόν την επόμενη Τετάρτη στις 23. Θα προτείνουμε λοιπόν αυτό το ποσό μέσω του ίδιου μείγματο επαναπρογραμματισμού και νέου χρήματος, όπως είχαμε προτείνει και πέρυσι. Δεν θέλω να προδικάσω την απόφαση της Κομισιόν, γιατί πρέπει να την πάρει, ακόμα δεν την έχει πάρει, αλλά αυτό προβλέπουμε να γίνει. Σε ό,τι αφορά την Ιεμένη, έγινε μια διάσκεψη του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, στις 3 Απριλίου, η Σουηδία και η Ελβετία ήταν συνδιοργανώτριες χώρες ως πήμα μιας ε, συνολικής δέσμευσης ύψους 2 ε, δισεκατομμυρίων δολαρίων έτσι, που έγιναν σε αυτή τη διάσκεψη. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε να δώσει το 2018 107 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό που αποτελείται από 37 εκατομμύρια από την ανθρωπιστική βοήθεια, το ΕΚΟ, αυτό ανταποκρίνεται στο αρχικό ποσό για την Ιεμένη στα πλαίσια του ανθρωπιστικού εργαλείου. Εν το συζητήσαμε και υιοθετήσατε μία μεταφορά για να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτό το ποσό για την Ιεμένη από το αποθεματικό κατεπίγουσα βοήθεια. Αυτό δεν ήταν τμήμα τη ε, δέσμε που είχαμε αναλάβει στι αρχέ του Απριλίου, γιατί δεν είχε ληφθεί τότε αυτή η απόφαση για τη μεταφορά, αλλά αυτή η ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την Ιεμένη, θα πάει στην Ιεμένη. Καταρχά, λοιπόν, έχουμε τα 37 εκατομμύρια από την ανθρωπιστική βοήθεια. Επίση, έχουμε 66 εκατομμύρια από το DCI, από την αναπτυξιακή βοήθεια. Και το τρίτο στοιχείο είναι 5 εκατομμύρια από το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Από το DCI, από την αναπτυξιακή βοήθεια και το τρίτο στοιχείο είναι 5 εκατομμύρια από το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Αυτές οι τρεις συνιστώσεις μας δίνουν 107,5 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση για τους πρόσφυγες, για την Τουρκία, το μηχανισμό αυτό χρηματοδότησης. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα 28 κράτη-μέλη είναι έτοιμα να φτάσουν σε ομόφωνη συμφωνία, περίπου έτοιμα, ότι οι, οι διμερείς, όμως, ότι οι διμερείς συνεισφορές των κρατών μελών θα πρέπει να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο. Η επίσημη συμφωνία δεν έχει ε, ληφθεί ακόμα, γιατί υπάρχει μία χώρα η οποία δεν έχει κυβέρνηση και περιμένουμε την επίσημη συμφωνία αυτής της χώρας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε πολύ σύντομα ε, ομόφωνη συμφωνία για το θέμα του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τους πρόσφυγες για την ε, Τουρκία. Από πλευρά Συμβουλίου, αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 2 δισεκατομμύρια θα πρέπει να τα βρούμε από τον ενωσιακό προπολογισμό. Τελευταίο ενημερωτικό σημείο για τον επόμενο σχέδιο, για το επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού την επόμενη Τετάρτη για το 19 θα υιοθετήσουμε και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3 για το 18, που θα έχει την πρόταση για τη χρηματοδότηση του κομματιού του FRT για το 2018 τμήμα των 3 δισεκατομμυρίων και 31 Μαΐου η Κομισιόν θα υιοθετήσει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμό 4, που είναι ένα μικρό ποσό για τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης, που αφορούν τις πλημμύρες κυρίως στη Λετωνία, Λιθουανία και Πολωνία. Το επόμενο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού όπως κάθε χρόνο, είναι η προσαρμογή των εσόδων και η επικαιροποίηση των ιδίων πόρων που θα είναι ο διεθνωτικός προπολογισμός παριθμών 5. Δεν ξέρω πότε θα υιοθετηθεί ακόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γιατί... Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τώρα ο κ. Μυροσάνο, ο γενικός μας συζητητής, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που είσαστε και εσείς μαζί μας σήμερα, γιατί ακριβώς τέτοιου είδους ε, δουλειά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε από κοινού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που είσαστε και εσείς μαζί μας σήμερα, γιατί ακριβώς τέτοιου είδους ε, δουλειά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε από κοινού σε όλα τα δημοσιονομικά έτη. Αυτό ήταν ε, και ο σκοπός μας στις αρχές του έτους, να υπάρχει τακτική ανταλλαγή απόψεων και να φροντίσουμε η εκτέλεση του προϋπολογισμού να μην ε, μας απογοητεύσει.